Μετά από την παρέτηση του κυρίου Μάλτιν Σούλτς, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να τη χειρεύει θέτη του από τις 17 Φεβρουαρίου 2017 και ε, ε, ενημερώνει και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Από